που θα εισηχθεί από τον Απρίλιο και μετά. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις ε, ψηφίσματος. Κλείνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο, Τετάρτη, στις 12. Μετά τα αυτά, κλείνω εδώ τη συζήτηση. Και σταματά εδώ η συνεδρία της Ολομέλειας. Αύριο, 11 Μαρτίου, 9 το πρωί, ξαναρχίζει η Ολομέλεια. Δημοσιεύθηκε και στο website του Κοινοβουλίου ε, η μερίσια διάταξη. Σταματά